Και τώρα θα περάσουμε σε επεξηγήσεις ψήφου. Πρώτο για την έκθεση Λουκαντράουι. Ο κύριος Γκόλνις. Κύριε Γκόλνις. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης του κυρίου Καντράουι για το καθεστώς αμοιβή των ε, στελεχών των επιχειρήσεων που είναι εντεταγμένε στο χρηματιστήριο. Στη Γαλλία όλοι αυτοί συνήθως προέρχονται από μεγάλε, από ε, τα διάφορα υπουργεία ε, και συσσωρεύουν με πραγματικά αναξιοπρεπή τρόπο τις ώρες παρουσίας στα υποτιθέμενα συμβούλια και λαμβάνουν διάφορα πρίμα τη στιγμή που φεύγουν, χαίρουν αυτού που αποκαλούμε χρυσή χειραψία. Πρόκειται για πράγματα που γίνονται εκτός ελέγχου με πραγματικές σχέσεις που έχουν να κάνουν με επιχειρήσεις των οποίων οι μέτοχοι όπως και οι υπάλληλοι υποφέρουν από την έλλειψη ικανότητας. Αυτή η κατάσταση είναι πραγματικά αβάσταχτη, δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί, πρέπει να πάψει ε, πηγόντως, διότι αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, η οικονομία της αγοράς και ο καπιταλισμός θα χάσουν κάθε εξοπιστία. Uh, next, Mr. Hannan, please. Hannan, Κυρία Πρόεδρε, εμείς θέλουμε να ρυθμίσουμε τους όρους και προποθέσει για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. Ορισμένοι βουλευτές θα θυμούνται ότι προέρχονται από χώρες που αυτό ήταν υπόθεση του κράτους. Ακόμα και στη δική μας χώρα, στη ε, δεκαετία του 70, με καταστροφικές συνέπειες. Δεν είναι υπόθεση των, των κυβερνήσεων να αποφασίζουν τι ε, ποια θα είναι η αμοιβή μου. Αν εγώ θέλω να δουλέψω για εσάς Πρόεδρε και είμαι ικανοποιημένος με τους όρους του σύμβαση μου, είναι δική μου υπόθεση και όχι κρατική υπόθεση. Οι κυβερνήσεις θέλουν να μειχθούν στις υποθέσεις των τραπεζών. Είναι ένα είδος ε, να υπάρξει μια ε, βαλβίδα ασφαλείας η οποία θα λειτουργήσει ώστε να φύγει ο θυμός που επικρατεί. Πολλοί, πολλοί επίσης ενέργησαν για να βοηθήσουν διάφορες από τους πλουσιότερους ανθρώπους να ξεφύγουν από την πλήρη κατάρρευση. Ακόμα και αν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει μέσω των σωστών δημοκρατικών εθνικών μηχανισμών των κρατών μελών και όχι να επιβληθούν από τις Βρυξέλλες. Ο κύριος Καμάλα. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που σας βλέπω για μια ακόμη φορά να προεδρεύετε. Προφανώς η επίδοση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και θα πρέπει να οργιζόμεθα από τα στελέχη των μεγάλων τραπεζών που πολλές φορές είναι στην πορεία της πτώχευσης, αυξάνουν τα χρέη τους και όμως αυτοί πληρώνονται άψογα. Θα πρέπει όμως επίσης να γνωρίζουμε και τις συνέπειες αυτών των ρυθμίσεων και πολλές φορές δεν το γνωρίζουμε. Αν πράγματι εμείς επηρεάσουμε και ρυθμίσουμε το κειμενόμενο τμήμα των αμοιβών και τα λεγόμενα μπόντους, θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι τράπεζες αυτές. Προφανώς θα αυξήσουν τον βασικό μισθό και θα μειώσουν την κειμενόμενη και εξαρτώμενη από τις επιδόσεις εν αμοιβή τους τελέχους τους Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να μελετήσουμε προσεκτικά τις απρόβλεπτες συνέπειες που θα έχει η απόφασή μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στόχος του κανονισμού είναι να ρυθμίσει την είσοδο στις αγορές νέων καινοτόμων τροφίμων και τροφίμων από τις τρίτες χώρες. Εισάγονται νόμοι για την ετικετοθεσία και την εμπορία των νέων αυτών προϊόντων τροφίμων. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης είδαμε ότι το Κοινοβούλιο προσπάθησε να δώσει εγγυήσει στην προστασία της υγείας, της ανθρώπινης ζωής, της ευημερία των ζώων, του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. Το Συμβούλιο όμως έλαβε υπόψη του τμήμα μόνο αυτών των στοιχείων κατά τη διάρκεια της πρώτης αναγνώσεως. Συνεπώς, δεν ελήφθησαν υπόψη από το Συμβούλιο ορισμένε απόψει μας και γι' αυτό τις καταθέτουμε εκ νέου στο Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα σχετικά με τα κλωνοποιημένα τρόφιμα και ε, σε σχέση με τα τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και για τις ζωοτροφές μέσω των τροπολογιών μας εισάγουμε τις απαραίτητες εγγυήσει σχετικά ε, με την προέλευση και τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται κατά την εκτροφή των ζώων. Καλενόφσκι. Pani Przewodnicząca, miesiąc temu głosowaliśmy nad dokładnym i jednolitym e, znakowaniem żywności, aby zapewnić konsumentom dostęp. Σχετικά με την ετικετοθεσία Νομίζω ότι απαιτούνται ε, περισσότερες πληροφορίες για το τι περιέχει ένα τρόφιμο. Αν πράγματι εμείς ε, ενδιαφερόμεθα για την υγεία των καταναλωτών, <clears throat> δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να δεχθούμε να κυκλοφορήσουν προϊόντα τα οποία έχουν ζωική προέλευση από ζώα που έχουν κλωνοποιηθεί. Θέλουμε προϊόντα γεμάτα υγεία για τους καταναλωτές μας και δεν θα πρέπει εμείς να εγκαταλείψουμε τα τρόφιμα τα οποία γνωρίζουμε ότι δεν είναι επικίνδυνα και αντίθετα να πειραματιστούμε με επικίνδυνα τρόφιμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η τεχνολογία επιβάλλει, θα έλεγα, και στα διάφορα κράτη, σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, να προσαρμόζει συνεχώς τους κανονισμούς και τις νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες έχουν σαν στόχο να προστατεύσουν την υγεία και την ποιότητα του τρόφιμου. Αυτό θα πρέπει να γίνεται και σε σχέση με τους κανόνες της ελεύθερης κυκλοφορίας των τροφίμων, εφόσον βέβαια τα τρόφιμα αυτά είναι ασφαλή. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και για μια νομοθετική θα έλεγα δραστηριότητα αποτελεσματική. Οι απόψεις τις οποίες υιοθετήσαμε σήμερα σύμφωνα με τις προτάσεις του Συμβουλίου προτείνουν να καταγραφούν στο συγκεκριμένο κατάλογο όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία εμπεριέχουν καινοτόμα χαρακτηριστικά και αυτό με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι σαφής η απουσία προσθέτων και τεχνολογιών που τροποποιούν γενετικά τη σύνθεση των προϊόντων αυτών και που προέρχονται πολλές φορές από τρίτες χώρες, ξένες χώρες, ξένες προς την ε, ενιαία αγορά. Γι' αυτό λοιπόν και στα πλαίσια του παρόντος νομοθετικού πλαισίου είμαστε ικανοποιημένοι από τα μέτρα τα οποία λήφθησαν. Ε, Κυρία Πρόεδρε, διαπιστώνω καταρχήν ότι δεν υπάρχουν οικονομικές ε, απαιτήσεις, απαιτήσεις για τη χρήση κρέατος από κλωνοποιημένα ζώα. Δεύτερον, οι, οι κίνδυνοι δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως για τέτοια τρόφιμα και δεν είναι συμβατή αυτή η διαδικασία με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Γι' αυτό η κλωνοποίηση ζώων για την παραγωγή τροφίμων είναι, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι αναμένει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση εκ μέρους μας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση. Οι ταχύες επιστημονικές εξελίξεις έχουν διευκολύνει την παραγωγή καινοτόμων τροφίμων. Ωστόσο, τα που που παράγονται με, στη βάση γενετικά τροποποιημένων ζώων δημιουργούν πάρα πολλέ ανησυχίε όσον αφορά τι επιπτώσει αυτών των ροφήμων στην ε, δημόσια υγεία. Οι επιστημονικέ και τεχνικέ εξελίξει είναι ωστόσο θα πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα ασφαλεία και θα πρέπει, δεν θα πρέπει να αφήνουν κανένα περιθώριο ε, υποψίες ή αμφιβολιών όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου στις αγορές. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν επαρκείς πληροφορίες για τέτοιου είδους τρόφιμα. Uh, Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα και ρετήσω από την Επιτροπή να υποβάλει την πρόταση για την κλωνοποίηση των ζώων που uh, απαγορεύει αυτά τα ζώα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν το θέλουν οι καταναλωτέ και γιατί του ενδιαφέρει η ευημερία των ζώων. Η Επιτροπή είπε ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη κλωνοποίηση για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του τροφίμων στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι είναι κάτι κακό για τα ζώα. Η κλωνοποίηση είναι χρονοβόρο και δαπανηρή. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχιστούν οι έρευνε και να ενθαρρύνουμε την Επιτροπή και την ΕΦΣΑ να καταλήξουν σωλημένε καινοτομίε και να αναπτύξουν τη τεχνολογία ό,τι αφορά αφορά τις υπόλοιπες της Ένα σημαντικό θέμα είναι ότι οι διάφορες δοκιμές δεν μπορούν να δείξουν διαφορά μεταξύ του κλωνοποιημένου και μη κλωνοποιημένου κρέματος. Συνεπώς δεν μπορούμε να ενημερώσουμε το καταναλωτή και να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να, να επιλέγουν ελεύθερα όπως εξάλλου έχουν δικαίωμα να κάνουν. Κυρία ψηφίσαμε υπέρ τη έκθεση, γιατί δεν έχουμε επιβαρκεί πληροφορίες σε ό,τι αφορά την επίπτωση των τεχνολογιών στα είδη διατροφή. Υπάρχει απαγόρευση της κλωνοποίηση και πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό, γιατί η έρευνα μας επέτρεψε να διαπιστώσουμε ότι προκύπτουν ασθένειες, παραμορφώσεις, διαμαρτίες αναποτέλεσμα της κλωνοποίησης. Συνεπώ επέρχονται αλλαγές σε κυταρικό επίπεδο και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουμε ολοκληρωμένα κλινικά στοιχεία όπω γίνεται για τα φάρμακα. Είναι απαραίτητο να υπάρξει απαραίτητη ταξινόμηση και για το λόγο αυτό θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η νανοτεχνολογία θα πρέπει να συμβάλλει έτσι ώστε να γνωρίζουν οι καταναλωτέ τι αγοράζουν. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα κατά τροφίμων που παράγονται από κλωνοποιημένα ζώα στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ τη πρακτική χρήση και τη επιστημονική έρευνα σε ό,τι αφορά τρόφιμα που προέρχονται ή διατροφή που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών είναι κατά του κλωνοποιημένου κρέατος και συνεπώς εμείς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτή τη γνώμη. Η ποιότητα αυτού του κλωνοποιημενου κρέατο. και συνεπω εμεί θα πρεπει είναι αφισβητήσιμη γιατί δεν γνωρίζουμε την επίπτωση που μπορεί να έχει στην ανθρώπινη υγεία. Μια άλλη πτυχή του θέματος είναι η ηθική. Σήμερα στέλνουμε ένα μήνυμα και λέμε ότι είμαστε κατά της πόλης προϊόντων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και λέμε στην Επιτροπή να υποβάλει μια νομοθετική πρόταση για αυτό το θέμα. Ο κύριος Στάκουλα. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω ότι υπερψήφισα την, τον, την κατάργηση του κρέατος που προέρχεται από κλωνοποιημένα ζώα. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να υπερψηφιστούμε μια υγιή ζωή δεν πρόκειται μόνο για το κέρδος, πρόκειται και για την ευημερία των ζώων καθώς και την υγεία των ανθρώπων. Θα πρέπει να έχουμε καθαρά τρόφιμα για όλους τους καταναλωτές. Και θα πρέπει, δεν θα πρέπει οι δυνάμεις της αγοράς να καθορίζουν την ε, υγεία των καταναλωτών. Είναι σημαντικό να έχουμε επαρκείς πληροφορίες και έρευνες για το κλωνοποιημένο κρέας, για το κρέας παρά για τα αποκλεινοποιημένα ζώα. Και υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι οι επιπτώσεις στην υγεία δεν είναι θετικές και είναι δυνατόν να υπάρχουν και νόσοι που ανάγονται στη χρήση τέτοιων τροφίμων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πράδα, Είναι ε, μεγάλη χαρά που μπορώ να σας ε, αποκαλέσω αξιότιμοι φίλοι σαν ε, ως αποτέλεσμα των τελευταίων εξελίξεων. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και τους άλλους φιλελεύθερους βουλευτές για το ρόλο που παίξατε για την νομοθεσία αυτή που εν μέρει έχει ε, αναβληθεί όσον αφορά τη δημιουργία νέων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η πλειοψηφία των ε, οικονομικών υπηρεσιών επικεντρώνεται στην πόλη του Λονδίνου. Πρόεδρος ε, Διακόπτη. Κύριε Χάμον, θα πρέπει να αναφερθείτε στην έκθεση Λιωτάρ. Για... Σε αυτήν αναφέρονται επεξηγήσεις ψήφου. Θα περάσουμε στην έκθεση Κρέμερ. Κύριος Καλενάσκη. Pani Przewodnicząca, dziękuję bardzo. Trzeba wykorzystać wszelkie Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όλες τις τεχνολογίες που έχουμε στη διάθεσή μας για τη μείωση των εκπομπών από τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις που πήραμε σήμερα προωθούν αυτές τις νέες τεχνολογίες, οδηγούν στο streamlining, όπως λέμε, και στον εναρμονισμό των ομοθετικών ρυθμίσεων. <clears throat> Θα πρέπει να αποφύγουμε περαιτέρω γραφειοκρατικές περιπλοκές, σεβόμενοι τα μέσα τα οποία παρέχει η αγορά, και δεν θα πρέπει προσπαθώντας να κάνουμε το καλύτερο να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το πρόβλημα τη ρήπανση μα επιτρέπει θεσμικά να είμαστε παρόντε και να αντιμετωπίζουμε με σαφήνεια το πρόβλημα των ε, βιομηχανικών εκπομπών. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική για να μπορέσουν να ζήσουν και οι υπερχόμενες γενναίες. Η προστασία της ατμόσφαιρας, του εδάφους, των υδάτων επιβάλλει σήμερα σε όλα τα θεσμικά επίπεδα την τελειοποίηση στρατηγικών ελέγχου και περιορισμού των ε, ρήπων έτσι ώστε να μπορέσει να επανεξεταστεί η αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον. Αυτό δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να υιοθετήσουμε ιδιαίτερα δίσκαμπτη στάση σε ό,τι αφορά την βιομηχανία. Και σε μια στιγμή οικονομικής κρίσης υπάρχει ο κίνδυνος να καταβάλουν ένα υψηλότατο τίμημα. Συμφωνώ με την έκθεση, αλλά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την ανάγκη που υπάρχει να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και να λάβουμε υπόψη μας στόχους, όπου, ε, στόχους που θα συμπεριλαμβάνουν όλες τις χώρες Ο κύριος Βαρθολούτσι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόκληση για την πρόληψη της ρήπαση σε σχέση με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις είναι ένα ιδιαίτερα επίκαιρο πρόβλημα που αφορά διάφορους τομείς μεταξύ των οποίων την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία των πολιτών και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η συγκεκριμένη οδηγία από την άποψη μιας σφαιρικής προσέγγισης ό,τι αφορά το σημαντικό αυτό θέμα ε, ακολούθησε το στόχο εφαρμογής καλύτερων τεχνικών που θα οδηγήσουν στον έλεγχο των εκπομπών και στη δημιουργία προτύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να υπάρξουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις που μπορούν να προστατεύσουν το περιβάλλον που πολύ, ενώ πολύ συχνά υπάρχει ο κίνδυνο συμβιβασμού. Σε όλα αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανάγκη και των βιομηχανιών μας να μην χάσουν τον απαραίτητο ανταγωνισμό που θα τους, ανταγωνιστικότητα που θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν τις διάφορες προκλήσεις. Χρειάζεται βεβαίως πολιτική δέσμευση και βούληση. Θα πρέπει να υπάρξει διαμεσολάβηση, χάρη στην οποία θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μια συμφωνία με την ευκαιρία του τρίτου ε, τριμερούς διαλόγου. Θα ήθελα για τον λόγο αυτό να υποστηρίξω αυτή την έκθεση. Ο κύριος Μετσάρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα δεν μπορεί κανείς, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το περιβάλλον με αποσπασμητικές ενέργειες. Γι' αυτό και έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την περίπτωση του IPCC και όπου ένας, καλύπτεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός βιομηχανικών μονάδων γιατί ανάμεσα σε αυτές τις βιομηχανικές μονάδες υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι ε, πρωταγωνιστής θα έλεγα στην μόλυνση του περιβάλλοντος. Αν θέλουμε να πετύχουμε όμως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε καλύτερα τα νομικά τουλάχιστον μέσα τα οποία θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν σωστά ό,τι περιλαμβάνεται στα έγγραφα αναφοράς είναι σαφές ότι απαιτούνται εκατότατα επίπεδα στα πλαίσια του ελέγχου των εκπομπών. Περνάμε στην έκθεση Χάση. Κύριος Καλενόφσκι πάλι. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, lasy obok fundamentalnych funkcji, jakie pełnią dla środowiska, będąc najbardziej trwałe. Τα δάση παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για το περιβάλλον. Είναι από τα πιο διαρκή χρονικά οικολογικά συστήματα τα οποία διαμορφώνουν το τοπίο πάνω στη γη. Και φυσικά παίζουν και πολύ σημαντικό οικονομικό ρόλο στις περιοχές της Υπέθρου. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε ε, την αποψήλωση των δασών και να βοηθήσουμε την διατήρηση της ποικιλότητα ε, του, ε, της χλωρίδας και της πανίδας στις περιοχές της δασικές. Υπήρξαν σοβαρά προβλήματα σε ορισμένε δασικέ εκτάσει την προηγούμενη εβδομάδα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη λόγω των πλημμυρών. Your. Χαιρετίζω πάρα πολύ που η Επιτροπή θέλει να καταπολεμήσει την παράνομη υλοτόμηση. Εν ώψη των δραματικών επιπτώσεων τη παράνομη υλοτόμηση και τη αποψήλωση των δασών, κάτι τέτοιο είναι απολύτω αναγκαίο. Ωστόσο, ήταν απαραίτητο να υπάρξει ένα ισορροπημένο συμβιβασμό, ο οποίο να μην ε, θέτει μη αναγκαία εμπόδια στι βιομηχανίε ε, ξύλου. Νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα της αποψήλωσης των δασών. Ωστόσο υπάρχει ένα αθέμητο πλεονέκτημα του ανταγωνισμού το οποίο έχει δημιουργηθεί λόγω της παράνομης υλοτόμησης και με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται. Έτσι λοιπόν η ξυλία θα μπορεί να προέρχεται μόνο από επιτρεπόμενες πηγές. Aikomus laittomien ο στόχος της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης είναι να καταπολεμήσει την παράνομη υλοτόμηση παράνομα προϊόντα ξυλίας. Θεωρώ ότι είναι φταίος αυτός ο στόχος, γι' αυτό υπερψήφισα τον κανονισμό. Βεβαίως υπάρχουν κάποια προβλήματα στο επίπεδο της εφαρμογής όσον αφορά τους ε, παράνομους ε, παράγοντες στο τομέα αυτό, όσους εμπορεύονται δηλαδή παράνομη ξυλία θα πρέπει να σκεφτούμε ότι το μεγαλύτερο τμήμα της ε, ξυλίας προέρχεται από μη παράνομες ε, πηγές. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να θέτουμε μη αναγκαία εμπόδια στο εμπόριο. Ε, και στις ε, βιομηχανίες. Ναι μεν ε, ο στόχος είναι ευκταίος, αλλά θα, η χνηλασιμότητα της προέλευσης του ξύλου προσκρούει σε πολλά εμπόδια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε τελικά την τελευταία πηγή του ξύλου, σε όλη τη διαδικασία και δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε επιπλέον προβλήματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα έρθουμε στην έκθεση Sanchez ε, Ποσέδο. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μπορούμε να κατηγορήσουμε πολλούς για τα προβλήματα του πιστοτικού συστήματος. Μπορούμε να κατηγορήσουμε τις κυβερνήσεις που κράτησαν τα επιτόκια χαμηλά για πάρα πολλά χρόνια αλλά δεν νομίζω ότι θα διορθώσουν τίποτα οι προτάσεις αυτές. Είναι μια αντίδραση αποσπασματική και συναισθηματική ενάντια σε όσους εργάζονται στα χρηματοπιστωτικά. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει για κάποιες χώρες οι οποίες δεν έχουν μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα, αλλά η δική σας χώρα που είναι και δική μου συγκεντρώνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της δραστηριότητας αυτής που αφορά και τις κυβερνητικές λειτουργίες. Και νομίζω ότι σε επίπεδο χρηματοπιστωτικό θα έχουμε στη χώρα μου να ζήσουμε για μια ακόμη φορά μια νέα καταστροφική πολιτική αντίστοιχη με την κοινή πολιτική αλίας Κάποια, κάποια μέλη εδώ, επειδή είναι εναντίον του καπιταλισμού ή εναντίον του Λονδίνου γιατί μας ζηλεύουν, προφανώς θα υπερψηφίσουν τις ανόητες αυτές προτάσεις. Έκθεση Γκουλάρ. Ο κ. Αντωνιώτση έχει το λόγο για την έκθεση Γκουλάρ. Κύριε Αντωνιώτση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η παρούσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έδειξε το πόσο είναι αναγκαίο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα σύστημα οικονομικού ελέγχου που αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο για να μπορέσει να κρατήσει μακριά άλλες παρεμφερείς κρίσεις. Θεωρώ ότι η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συστημικό κίνδυνο είναι ο καλύτερος δρόμος για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την εσωτερική αγορά, για να εξασφαλίσουμε τη συνοχή των αποφάσεων και για να μπορέσουμε να ταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών που εδώ και πολύ καιρό αναμένουν την ε, ανάληψη συγκεκριμένων μέτρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ όλων αυτών των εκθέσεων που έχουν σχέση με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης και της έκθεσης του συναδέλφου Μαρκάιο. Η νομοθεσία για τα χρηματοπιστωτικά συστήματα έχει σκοπό την καλύτερη ρύθμιση της δράσης των ε, αγορών και στα μέτρα που αφορούν τα προβλήματα σε αυτό το τομέα. Αυτό είναι κάτι που απαιτείται για να αντιμετωπιστούν μελλοντικέ κρίσεις. Είναι σαφές ότι μια χρηματοπιστωτική αγορά που δεν ε, ρυθμίζεται καλά θα καταλήξει σε μια περαιτέρω ύφεση. Η χρηματοπιστωτική κρίση δημιούργησε πάρα πολύ σοβαρούς κινδύνους, οδήγησε σε μία αστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της εσωτερικής αγορά. Για να αποφύγουμε το φαύλο κύκλο τις ε, αγορές θα πρέπει να υιοθετήσουμε περισσότερο σωστούς καμισμού. Η εταίροι μας στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένε Πολιτείε έχουν λάβει τέτοια μέτρα. Ήρθε η ώρα να γίνει το ίδιο και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε περίπτωση που έχετε αφιβολία, συζητάμε την έκθεση Καρθία Μαργκάλο ή Μάρφυρ, ο επόμενος ομιλητής, κύριος Αντώνιος Σιέγγεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι υπέρ του να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, γιατί αυτό το εργαλείο θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει τα κανονιστικά κενά που εντοπίσαμε ότι υπάρχουν κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Κενά που εδώ και καιρό έχει εντεπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω κατέστησε σαφέ από ορισμένε εκθέσει που επιβλήθησαν σχετικά με αυτό το θέμα, ο συντονισμό και μόνο μεταξύ των αρχών ελέγχου, των οποίων ε, που κινούνται στα πλαίσια των χωρών μελών δεν είναι υπαρκή για τον έλεγχο αυτών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αντιλαμβάνονται την εσωτερική αγορά ως ένα χώρο ξέφραγο. Η δημιουργία αυτής της αρχής θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο σημαντικό βήμα για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παλώνε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτές οι ανεξάρτητες αρχές που θα είναι ισχυρές και θα έχουν τη δυνατότητα αντιβολής κυρώσεων είναι κάτι σημαντικό. Έχω όμως και ορισμένες αμφιβολίες, ορισμένα ερωτήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν γιατί οποιαδήποτε αναφορά σε επιβολή χρηματοπιστή θα πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν θα πρέπει η, να μεταφερθεί το κόστος, να μεταγυλήσει το κόστος στις μικρομεσαίες επιχείρησεις. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε ένα ενιαίο τραπεζικό σύστημα. Το Ιταλικό τραπεζικό σύστημα είναι σύστημα το οποίο βασίζεται σε υγιή κονδύλια και στις αποταμιεύσεις των πολιτών. Δεν είναι ένα σκερδοσκοπικό σύστημα όπως είναι, ε, διαπιστώθηκε σε άλλες χώρες. Πραγματικά ε, έχω όμω αμφιβολίες για ορισμένε χρηματοπιστωτικέ δράσεις που θα πρέπει να επαληθεύσουμε, ε, να ελέγξουμε κατά πόσο είναι κατάλληλες για ε, ιδιαίτερες συνθήκες. Θα πρέπει να ελέγξουμε τις αρμοδιότητες της τράπεζας σε ό,τι αφορά στις τελικές ομάδες και θα πρέπει να διευκρινίσουμε το, το ρόλο μεταξύ ε, της μικρο και μακρο, του μικρο και μακρο Ελπίζω η σημερινή ψηφοφορία να μας επιτρέψει να επιτύχουμε γρήγορα ένα συμβιβασμό με το Συμβούλιο. Ένα λεπτό θα πρέπει να είναι η παρέμβαση σα. Έκθεση Μακάρθη τώρα, Κύριο Στάκουλα. Κυρία Μακάρθη. Σήμερα υπεψήφισα την έκθεση Μακάρθη σεβόμενος την άποψη της πολιτικής μου ομάδας, αλλά υπάρχουν κάποια λαϊκιστικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν νομίζω ότι ανήκουν σε μια σωστή νομοθετική δραστηριότητα. Προφανώς δεν θα πρέπει οι τράπεζες να υποστηρίζονται συστηματικά από τους φορολογούμενους, αλλά αυτοί η πολύ αυστηροί κανονισμού, δεν είναι τέτοιου είδους έτσι ώστε να καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά πολύ περισσότερο από τις κεντρικές κυβερνήσεις των κρατών μελών. Αυτές οι κεντρικές τράπεζες ε, θα πρέπει να αποφασίζουν ε, αν κάτι είναι λογικό και πρέπει να ε, γίνει σεβαστό και κάτι είναι υπερβολικό και θα πρέπει να καταπολεμηθεί. Υπάρχουν στις προτάσεις Μακάρθη πάρα πολύ θετικά στοιχεία και σε σχέση με την αυτορύθμιση και νομίζω ότι οι τράπεζες μπορεί να μπορέσουν να δουλέψουν ε, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν για να αποφύγουμε παλιές κρίσεις. Ο κύριος Μαστέλα για την έκθεση Φερέιρα. Η πρόσφατη νομοθετική κρίση θέτει την αναγκαιότητα ε, παρέμβασης για να εγγυηθούμε την επιβιωσιμότητα και την αηφορία του συστήματος του χρηματοπιστωτικού. Βέβαια οι παρεμβάσεις και τα μέτρα θα έχουν τεράστιο κόστος και μπορεί να οδηγήσουν στο πάγωμα κάποιων χρηματοπιστωτικών αγορών, στη μείωση της χορήγησης πιστώσεων, σε αύξηση της ανεργίας και ε, γενικά σε μείωση των φορολογικών εσόδων. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Τα διάφορα μέσα και οι στρατηγικές Made in USA θέτουν ε, πολλές αμφιβολίες και δημιουργούν μια νομική αβεβαιότητα και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Παρ' όλα αυτά απαιτούνται σφαιρικές αποτελεσματικές λύσεις μέσω μιας ρύθμισης των διαδικασιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδείξει ότι είναι διαθέσιμη να πάρει μέρος σε ένα νέο προγραμματισμό, όχι μόνο στο εσωτερικό των 27 χωρών αλλά και σε διεθνές επίπεδο για το μέσο σταθερότητας η κυρία Ποδηματά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η κοινοβουλευτική μας ομάδα καταψήφισε σήμερα το ψήφισμα που αφορά τις αποφάσεις της 9ης Μαΐου για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής διευκόλυνσης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τον ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης παρά το γεγονό ότι θεωρούμε τι αποφάσει αυτέ εξαιρετικά θετικέ και σημαντικέ για την προστασία του ενιαίου νομίσματος και τη σταθερότητα τη ζώνη του ευρώ. θέλω να υπενθυμίσω με την ευκαιρία ότι το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πολύ καιρό πριν ζητούσε από το ευρωπαϊκό συμβούλιο να προχωρήσει προ την κατεύθυνση αυτή στέλνοντα ένα μήνυμα ενότητα και αλληλεγγύη προ τι αγορέ. πιστεύουμε όμω παράλληλα ότι την ίδια ετοιμότητα και αλληλεγγύη επέδειξε και η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα με την απόφασή τη για προσωρινή παρέμβαση στη δευτερογενή αγορά ομολόγων μια απόφαση που ήταν σε απόλυτη συμφωνία με το γενικότερο πνεύμα της απόφασης του συμβουλίου των υπουργών οικονομίας. δεν αντιλαμβανόμαστε λοιπόν και δεν συμμεριζόμαστε το πνεύμα της παραγράφου 14 με την οποία ασκείται κριτική στην ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα για την απόφασή της αυτή. σας ευχαριστώ πολύ piedāvātie Κύριε Πρόεδρε, οι μηχανισμοί σταθερότητας που προτείνονται εδώ, παρόλο που είναι κάπως καθυστερημένοι, μπορούν να προσφέρουν μια διευκόλυνση των χωρών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες. Αλλά δεν πρόκειται παρά μόνο για προσωρινά μέτρα. Η κρίση έδειξε πολύ ξεκάθαρα ότι πολλές χώρες, ιδιαίτερως εκείνες οι χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη, ε, αντιμετωπίζουν σημαντικότατα προβλήματα και δεν έχουν σωστό συντονισμό. Βεβαίως μπορούμε να συζητήσουμε όλες αυτές τις ιδέες μία διευκόλυνσης χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αλλά πριν δημιουργήσουμε ένα νέο θεσμικό όργανο θα πρέπει να ελέγξουμε το πώς ε, μπορούν να λειτουργήσουν οι παλιοί ε, θεσμοί. Θα πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου η σταθερότητα της Ευρωζώνης και των ε, μηχανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ε, αξιοπιστίας να υπονομεύονται. Ε, πολλές, όλες οι χώρες εκτίθενται στις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς. Για την Ισλανδία τώρα. Higgins. Εγώ ήμουνα κατά, γιατί ζητά τα δάνεια των Ισλανδικών τραπεζών να επιστραφούν χωρίς να διευκρινίζει ότι αυτό δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τον, καθη... μέσο ε, Ισλανδό πολίτη. Για να διασωθούν τα συμφέροντα δηλαδή των ε, καταθετών της Ολλανδίας και της Μεγάλης Βρετανίας, θα πρέπει να χρεωθούν οι φτωχοί Ισλανδοί οι οποίοι έχουν αρνηθεί κατά 80% σχεδόν με το δημοψήφισμά τους τις αποφάσεις αυτών που καταχράστηκαν, που έπαιξαν με το χρέος της χώρας τους και που δημιούργησαν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Επιβάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακόψουν τα κοινωνικά μέτρα εις βάρος των εργαζομένων χωρίς σε καμία περίπτωση ε, να, να ζητήσουν αντίστοιχα μέτρα εις βάρος των πλουσίων και των επιχειρήσεων και του χρηματοπιστωτικού τομέα και τελικά υιοθετούν ουσιαστικά τα μέτρα του κόμματος του κ. Χάναν απέναντί μου. Πρέπει να προειδοποιήσουμε λοιπόν το λαό της Ισλανδίας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της προκάλεσε την κρίση και δεν είναι φίλη της χώρας τους. Υπεψήφισα το ψήφισμα και θα ήθελα να υποστηρίξω να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία γρήγορα για να οδηγηθούμε πιθανώς σε μια χώρα νέο μέλος είναι μια ευρωπαϊκή χώρα με ισχυρή δημοκρατική κουλτούρα, ένα ισχυρό δημοκρατικό σύστημα και αναπτυγμένη οικονομία. Πράγματι είναι και πλέον η ώρα να διευρυνθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και προς περιοχές οι οποίες να εκπληρούν τα δημοκρατικά και οικονομικά κριτήρια. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να σταματήσει σήμερα και να μένουν χώρες όπως η Κροατία και άλλες χώρες της Βαλκανικής στη λίστα αναμονής. Και αργότερα ίσως ε, και η Γεωργία και η Λευκορωσία κτλ. Να πούμε ότι μέχρι τώρα η διεύρυνση ήταν μια επιτυχία και μετέτρεψε προς το καλύτερο στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Υπήρου το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο. Ας διασχίσουμε τον ωκεανό λοιπόν, ας εντάξουμε την Ισλανδία που θα είναι η πρώτη χώρα μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας που θα ενταχθεί. Ο κύριος Χάναν. Κύριε Πρόεδρε, μας συγκινεί ότι κάποιος θα ψηφίσει για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο, ε, πραγματικά το κοινοφούλιο φαίνεται πραγματικά να δείχνει μια ιδιαίτερα αισιόδοξη στάση. Και πραγματικά βλέπω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια χώρα που μεταμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια. Κανένα δεν μπορεί να αρνηθεί ότι πραγματικά πρόκειται για ένα μεγαλειώδες εγχείρημα. Έχουν φτάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο διαφύωσης. Εγώ βεβαίω, ε, είμαι δημοκράτη και δέχομαι την απόφαση των Ισλανδών. Αν θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα του υποστηρίξω. Δεν φαντάζομαι όμω ότι θα ψηφίσουν για να παραιτηθούν από τα πλεονεκτήματα ενό από τα μεγαλύτερα κοινοβούλια στον κόσμο, ότι θα απαρνηθούν την αυτονομία που βρίσκεται μέσα στο αίμα των Ισλανδών. Είναι ανεξάρτητοι αυτοί οι άνθρωποι και αυτό ε, είναι κάτι που οι μη Ισλανδοί δεν μπορούν να καταλάβουν και να εκτιμήσουν. εγώ ελπίζω ότι δεν θα ψηφίσουν για να παραδώσουν αυτή τη, για να παραιτηθούν αυτή τη δημοκρατία. Ναι, υπερψήφισα εδώ την έκθεση και δηλώνοντας ότι, λέγοντας ότι Χαίρομαι που η Επιτροπή έχει κάνει τόσο γρήγορα βήματα με την, ε, με την έναρξη και τη σύνεξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Η... Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί ο ρόλος και θέση της Ισλανδίας στον αρκτικό χώρο και θα ενισχυθεί και η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως η ίδια η Ισλανδία θα αποφασίσει κατά πώς θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια δημοκρατία, δημοκρατική χώρα η Ισλανδία αλλά βεβαίως στις διαπραγματεύσεις θα υπάρξουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική, την πολιτική γεωργίας και επίσης το εμπορικό κυνήγι των φαλενών και η εμπορία των προϊόντων από το κρέας φάλενας. Ε, ξέρουμε τι γίνεται στην Ιαπωνία και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβληματιστεί σχέση με το πώς θα συνεχίσει την πολιτική της στο επίπεδο αυτό. Διακόπτουμε μέχρι τις 3 το μεσημέρι.